Ε, της, των εξελίξεων και της μίας περτέρου προόδου για αυτό το σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση έχει περαταθεί και η ψηφοφορία όπως και για τα άλλα θέματα θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Ε, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Βέσφαλ για τη δημογραφική αλλαγή και τις συνέπειές της για την πολιτική συνοχής. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Βέσφαλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η δημογραφική αλλαγή συμπεριλαμβάνει μεταξύ των σημαντικών θεμάτων αυτής της εποχής. Στη Γερμανία κάθε δεύτερο κορίτσι το οποίο γεννιέται στη Γερμανία ε, θα, φτάσει στα 100 χρόνια. Η 30 η 13χρονη κόρη μου χαίρεται ε, για αυτό το γεγονός, αλλά θα πρέπει εδώ να αντιδράσει έγκαιρα και η πολιτική. Θα πρέπει να καταλήξει σε κάποιες ε, συνέπειες και να θέσει τις ε, πολιτικές προποθέσει πλαίσιο. Η έκθεσή μου, την οποία θα ψηφίσουμε αύριο, ασχολείται ακριβώς με αυτές τις επιπτώσεις και τις προϋποθέσεις πλαίσιο. Εδώ το ζητούμενο δεν είναι κοινωνικό όπως οι συντάξεις γιατί εδώ η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν είναι αρμόδια αλλά το ζητούμενο είναι ε, τι ε, πρέπει να πράξει η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής και πώ ε, θα πρέπει να διαμορφώσουμε μελλοντικά την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής ώστε να συμπεριλάβουμε τα σημαντικά θέματα και να τα προσεγγίσουμε. Συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφέρω τέσσερι τομεί που αναφέρουμε στην έκθεσή μας. Πρώτον, καταρχήν είναι αναγκαίο η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής να ενισχυθεί περισσότερο και να στραφεί σε φαινόμενα δημογραφικής μεταβολής. Στην Ευρωπαϊκή Στατική 2020 και στις νομοθετικές προτάσεις η δημογραφική μεταβολή παίζει έναν αρκετά σημαντικό ρόλο. Εδώ θα ε, και τώρα θα πρέπει να προσέξουμε για την εφαρμογή στην πράξη, ώστε το θέμα αυτό να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, ο τομέας υποδομές. Ε, χρειαζόμαστε ε, εδώ τα ε, δικαιοτοχή των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων στι κοινωνικέ δομέ για να αποκλείσουμε φαινόμενα αποκλεισμού. Για παράδειγμα, η πρόσβαση στα δημόσια κτίρια. Και παράλληλα, άλλε ομάδε, για παράδειγμα, οικογένειε με μικρά παιδιά ή οι ανάπηροι θα μπορέσουν να αποφεληθούν. Ταυτόχρονα, θα πρέπει ε, να προστατεύσουμε περιοχές και να τις καταστήσουμε πιο ελκυστικές που απειλούνται από την ε, έξοδο του πληθυσμού. Ε, τρίτον, ηλικιωμένοι και οικογένειες με παιδιά. Στις περιφέρειες της Ευρώπης ζουν όλο και περισσότερο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιδράσει έγκαιρη περιφερειακή πολιτική. Και εδώ συγκαταλέγεται για παράδειγμα για μένα η προώθηση σπιτιών στα οποία να διαβιούν περισσότερες γενιές αλλά επίσης ε, πρόθεση της υγείας. Ε, και όταν το ζητούμενο είναι να εμποδίσουμε την έξοδο του πληθυσμού, εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε για την ε, ημερήσια, ολοήμερη μάλλον, φροντίδα των παιδιών. Κρίμα που η πλειοψηφία της Επιτροπής τάχθηκε κατά του αιτήματο να παράσχεται δωρεάν φροντίδα, ολοήμερη φροντίδα των παιδιών. Εγώ θα ήθελα να είμαστε πιο θαραλέοι. Τέταρτον, ο τομέας απασχόληση, η καταπολέμηση της ανεργίας των ε, γυναικών και νέων θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Έχουμε μια γενιά νέων ε, γυναικών που έχουν την καλύτερη δυνατή κατάρτιση. Εάν αυτές οι γυναίκες δεν έχουν καμία ευκαιρία, με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουμε ένα έλλειμμα όσον αφορά τις ε, ε, το ειδικευμένο δυναμικό. Από την άλλη γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να. ότι πολύ περισσότερο την εμπειρία των ηλικιωμένων ή μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ε, περιφερειακές υποδομές. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει

Ε, ορισμένοι μεγάλες ορισμένες δεξιοδοτήθηκαν ε, κατά τη διάρκεια αυτής της, ε, του έργου. Ελπίζω να υπερψηφιστεί αύριο με πλατιά πλειοψηφία η έκθεση στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δημογραφική αλλαγή οφείλεται σε δύο αιτίες. ζουν όλο ένα και περισσότερα χρόνια οι άνθρωποι και γεννιούνται όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Σε αυτή την έκθεση εξετάζουμε τις δυνατότητες ενίσχυσης ε, της γεννητικότητας Υπάρχουν μέτρα που καταλύουν οικογένειες, ε, ποσοστώσεις για την απασχόληση των γυναικών. Όμως ε, οι γυναίκες ε, θα πρέπει να ανταμείβονται για την οικιακή τους εργασία, για την ανατροφή των παιδιών, την περίθαλψη άλλων μελών της οικογένειάς τους. Πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίσει την μη αμοιβόμενη εργασία και αυτό ε, να συνεπάγεται και εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η δημογραφική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα γεγονό και έχει αναδείξει σε βασική προτεραιότητα η προσαρμογή σε αυτή την αλλαγή. Αυτό οφείλεται σε χαμηλά ποσοστά γεννητικότητα, σε γέννηση του πληθυσμού, με μεταναστευτικέ ροέ, με μετακίνηση των πληθυσμών από την ύπεθρο προ τι πόλει. Όλε αυτέ οι αλλαγέ δημιουργούν νέε προκλήσει αλλά και ευκαιρίε. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει και να εκμεταλλευτούμε αυτέ τι ευκαιρίε. Ε, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη τα διαρθρωτικά ταμεία για να εκπονήσουν στρατηγικέ ε, για διαρθρωτικέ αλλαγέ που χρειάζονται. Σήμερα ε, στα κράτη-μέλη έχουμε τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή και κυρίω έχουμε στοιχεία κατά περιοχή. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για επαναπροσανατολισμό των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, ώστε να στηριχθούν οι γυναίκε που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επίσης, η φροντίδα των ελικιωμένων στην Ιρλανδία και αλλού θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Πρέντεγκαστ. Ο κύριος Μπάτιν τώρα. Η δημογραφία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ε, που κρύβει μεγάλες ιστορικές εξελίξεις ε, καθώς και ε, ιστορίες δημογραφικές που δεν έχουν ε, υποθεί ακόμα. Έχουμε μια ε, δημογραφική έκρηξη που δεν αναφέρεται στα ΜΜΕ. Όταν το 1997 ο Τόνι Μπλερ έγινε πρωθυπουργός, ήμασταν 58 εκατομμύρια. Σήμερα φτάσαμε στα 62,4 εκατομμύρια και με βάση τις σημερινές τάσεις θα ξεπεράσουμε τα 70 εκατομμύρια μέχρι το 2030 και εν συνεχεία θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ε, οι ειδικοί ε, υπογρα... Ε, λένε ότι αυτή η υπερβολική αύξηση οφείλεται στους μετανάστες και στις γεννήσεις των μεταναστών. Ε, κάνα πρόβλημα να υπάρχει μια μικρή ε, βιώσιμη μετανάστευση. Αλλά εμείς προσθέτουμε ένα εκατομμύριο ε, νέα άτομα κάθε 4-5 χρόνια. Ξεπερνάμε την ε, ε, Κίνα, την Ιαπωνία κτλ. Ε, αν μπορούσαμε χάρη στον πληθυσμό μας θα είχαμε καταλάβει την Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στη μεταναστευτική μας πολιτική. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή κοινωνία, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν πολλές δημογραφικές προκλήσεις ε, και την επόμενη δεκαετία θα είναι όλο και πιο έντονες. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής ε, είναι καλό, αλλά λόγω του χαμηλού ποσοστό γεννήσεων δεν αναιώνεται ο πληθυσμός. Ε, θα δημιουργήσει προβλήματα στα συνταξιοδοτικά, στο σύστημα υγείας και στην διαγενειακή αλληλεγγύη. Ε, μου κάνει εντύπωση που οι συντάχτες ε, δεν μιλάνε για όλα αυτά τα θέματα, δεν μιλάνε για την αρχική πυρηνική οικογένεια, τον πατέρα και τη μητέρα, γιατί από αυτό το κύτταρο προέρχονται τα παιδιά ε, σε αντιδιαστολή με τις μονογονικές οικογένειες κτλ. Ε, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια συζήτηση για τις δημογραφικές αλλαγές και τις νέες τάσεις ε, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα της ε, πολιτικής συνοχής με βάση τους δείχτες που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Κύριε Μορκουνάιτεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή έκθεση ε, για την επικοδομητική δουλειά που έκανε. Ήμουνα σκιώδης εισηγητής. Ο πληθυσμός γυράσκει στην Ευρώπη. Η Κομισιόν μιλάει για τη σημασία των δημογραφικών αλλαγών, για τις απειλές και τις δυνατότητε που δημιουργούν οι νέες τάσεις. Στο, ε, περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, τα κράτη-μέλη ξόδεψαν το 8,5 των ε, κονδυλίων των διαφορετικών ταμείων και η περιφερειακή πολιτική είναι το πρώτο εργαλείο ε, για να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικέ αλλαγές. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία. Ε, πρέπει να υποστηρίξουμε τι τοπικέ κοινότητε ε, όταν υιοθετούν αποφάσει για την πολιτική συνοχή. Το θέμα αυτό είναι σφαιρικό, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία. Πρέπει να δούμε και θέματα που απασχολούν την νεότητα και τις οικογένειες μην ξεχνάτε ότι τα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, αποτελεσματικά. Επίσης, ε, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τα συντοξιοδοτικά συστήματα τα οποία δημιουργήθηκαν όταν δημογραφικές τάσεις ήταν τελείως διαφορετικές από τις σημερινές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντανακλά την ε, πραγματικότητα, την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό κάνουμε και καλωσορίζουμε την έκθεση της ε, ε, κυρία Westphal, ε, μειώνεται ο αριθμός ε, γεννήσεων, γυράζει και ο πληθυσμός. Ναι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν δημογραφικές αλλαγές και άρα πρέπει να κάνουμε κάτι, να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση. Χρειάζονται πρωτοβουλίες εθνικές, αλλά και συντονισμός. Η περιφερειακή πολιτική είναι βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών και άρα Υποστηρίζουμε την τροποποίησή τη διαρθρωτική πολιτική τη Ένωση. Επίση, υποστηρίζουμε τη βοήθεια προ του ηλικιωμένου την ενίσχυση της γενετικότητας, τη διαγενειακή αλληλεγγύη, την ε, τους νέους, όσους βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και τους ηλικιωμένους. Ε, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στις πιο ευπαθείς ομάδες, οι γυναίκες, οι άνεργοι, οι φτωχοί, οι μετανάστες, οι ηλικιωμένοι. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει η πολιτική που ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε και ο κύριο Σικέρσκη ο τελευταίος ομιλητής για το Catch the Eye. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες και πολλές περιφέρειες. Έχουμε χαμηλά ποσοστά γεννητικότητα στην Ευρώπη. Από την άλλη έχουμε μεγάλη, πολλή μετανάστευση, ιδιαίτερα των νέων. Ε, οι νέοι πηγαίνουν προς τις μεγάλες πετροπόλεις. Η συγγήτρια έχει την άποψη, η διορθωτική πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο εξόδου και αναφέρεται σε έξι θέματα. Θα ήθελα να αναφερθώ στα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στις προκλήσεις που επέρχονται με τη δημογραφική μεταβολή. Η κατανομή των διαρθρωτικών ε, κονδυλίων θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις δημογραφικές εξελίξεις. Πέρα από αυτό, η συγκήτρια λέει ότι υπάρχουν προκλήσεις τόσο για τις πόλεις όσο και για την Ήπεθρο. Βεβαίω θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, υπάρξει μια μαζική έξοδος του πληθυσμού και βεβαίως οι πόλεις θα πρέπει να είναι πιο ελκυστικέ. Χρειαζόμαστε υποδομέ φιλικές προς τα παιδιά ή τις οικογένειες. Χρειαζόμαστε μια βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών. Και ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγων ε, είναι η αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων γυναικών. Αλλά βεβαίως χρειαζόμαστε τι αντίστοιχες υποδομές. εργαζομενων γυναικων αλλα βεβαιως χρειαζομαστε τι αντιστοιχε υποδομε τωρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Ντάλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Ε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Westphal για αυτή την έκθεση. Η έκθεση αυτή είναι μια πολύτιμη συνεισφορά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναγνωρίζει και η έκθεση υπάρχουν βασικές αλλαγές ε, βασικές διαφορές ω προ τι δημογραφικές αλλαγέ που θα γνωρίζουν ε, χώρες και περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωση. Άρα ενιαία προσέγγιση δεν ε, συνιστά πανάκια, δεν αποτελεί λύση για όλους. Έχουμε ήδη δραστηριε σε πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης, εξυγχρονισμό των υποδομών στον τομέα της υγείας, βρεφονιπιακή σταθμή, εργατική στέγη, υποστήριξη για την οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση των μειονοτήτων και των μεταναστών. Έχουν αναλυφθεί δράσει τώρα. Ο στόχο μας είναι να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με το πακέτο για το Ταμείο συνοχή για την περίοδο 14-20 που ενέκρινε στις 6 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, βλέπουμε με ε, μια σειρά επενδύσεων που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε αυτές τι δημογραφικέ ε, αλλαγέ. Αυτό καλύπτει τα τρία ταμεία που συμπεριλαμβάνει το πακέτο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είμαστε υπέρ της χώρες προσέγγισης, υπέρ της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, υπέρ μεγαλύτερης ευελιξίας όπου χρειάζεται και υπέρ νέων ευκαιρίων, ούτως ώστε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε τις δημογραφικές αλλαγές. Αξιοπρεπής υγιής γύρανση είναι κάτι το κέριο για την κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γυράς και ο πληθυσμός και η Ένωση στον τομέα της ε, υγείας έχει αναλάβει δράσεις και με αυτές τις δράσεις έχει βελτιώσει κατά πολύ την πρόσβαση στι υπηρεσίες της υγείας. Τώρα εκπονούμε μια στρατηγική πλαίσιο για να καλύψουμε αυτά τα προαναφερθέντα τρία ταμεία συν το Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέτρου καθώς και το Ταμείο Αλίας. Το πλαίσιο αυτό θα ε, απηχεί ε, του τους βασικούς τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής και θα υποστηριχθούν οι στόχοι από δράσει αυτών των τριών ταμείων. Θα προσαρμοστούμε στι δημογραφικέ αλλαγέ και θα προσδιορίσουμε πώ θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία ε, ανάμεσα στα τρία αυτά ταμεία. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε την έκθεση Vesta, West ε, Lab και τώρα ξεκινάμε το τελευταίο σημείο την έκθεση Simon, κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.